αυξήσουμε και την ανθεκτικότητα των αναπτυσσόμενων χώρων και των αναπτυγμένων χώρων στις, ε, στην κλιματική αλλαγή, όπως ε, αναφέρθηκε και στη σχετική συνάντηση της τελευταίας εβδομάδας. Ε, σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο αναμένω να ακούσω με ενδιαφέρον του, της απόψης του Ειδικού Συμβούλου κ. Ντάβιν Ναμπάρο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και της ατζέντα 2030. Επιχαίρουμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε αυτή την προσέγγιση, αλλά και για να ακούσουμε ποιες, ποια είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Χαιρόμαστε λοιπόν που είσαστε σήμερα μαζί μας κύριε Ναμπάρο και αναμένουμε να ακούσουμε από εσάς πώς ακριβώς θα εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα στην πράξη τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Ναμπάρο. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μου τιμή και προνόμιο το γεγονός να μπορώ να παρίσταμαι σε αυτή την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και της Επιτροπής για το Περιβάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να εκφράσω τη βαθιά μου ευχαρίστηση για το γεγονός ότι η επίσκεψή μου εδώ σήμερα για να σας συναντήσω συμπίπτει με την ε, δημοσιοποίηση δύο ανακοινώσεων. Τα επόμενα βήματα για ένα αηφόρο ευρωπαϊκό μέλλον και ε, η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Ξέρετε, ήμουνα εδώ στις Βρυξέλλες στις αρχές αυτής της χρονιάς για να εστιάσω την προσοχή μου στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη πρόκειται να προχωρήσει πάνω στα θέματα της αηφόρου ανάπτυξης. Ακούγοντας τους επιτρόπους και τους ε, αξιωματούχους, σκέφτηκα ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο να είναι εφικτό. Αναφέρομαι στη δημοσιο... δημοσίευση αυτών των δύο ανακοινώσεων μαζί πριν τη λήξη του έτους. Και είναι πολύ καλό και ευτυχές το γεγονός ότι διαψεύστηκα στις προβλέψεις μου και ότι τελικά οι δύο ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν την ίδια ημέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έτσι στέλνει ένα χειρότατο μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο εξ ονόματος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι, συνάδελφοι, αυτό που πραγματικά μετρά είναι ακριβώς αυτό. Ε, ε, φόρος ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια έννοια, αλλά είναι και μια προσέγγιση. Ένας τρόπος προσέγγισης ε, που βασίζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και ξέρετε, τίθεται συχνά το ερώτημα, επιθυμεί η Ευρώπη να συνεχίσει να ηγείται στον τομέα αυτό. Ε, λοιπόν, η δημοσίευση δύο ανακοινώσεων ταυτοχρόνως αποτελεί ένα ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα ότι πράγματι υπάρχει ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει συγκεκριμένη θέση για τα πράγματα. Και θα αναφερθώ σε αυτά εντός ολοϊγού, κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια να σας πω για την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030. Είναι μια ατζέντα πολιτική η οποία εγκρίθηκε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο του 2015 μετά από δυόμιση χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων. Πολλοί από εμάς που είχαν εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις τότε με μεγάλη χαρά παρακολούθησαν την δημιουργία και τη γέννηση, αν θέλετε, της ατζέντα για το 2030, κυρίως χάρη στα εξή χαρακτηριστικά της. Πρώτον, είναι παγκόσμια, είναι οικουμενική, ισχύει για όλες τις χώρες, για όλες τις κοινότητες στον κόσμο μας. Δεύτερον, είναι μια διασυνδεδεμένη ατζέντα. Οι 17 στόχοι ε, εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν 17 τομείς της ανθρώπινης ύπαρξης, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλο. Και τρίτον, θα εφαρμοστεί με τρόπο ώστε κανείς να μην μένει πίσω. Τέταρτον, θα εφαρμοστεί με ενίο, με ολοκληρωμένο τρόπο και τέλος θα εφαρμοστεί, θα εφαρμοστεί μέσω εταιρικών σχέσεων πολυμερών και με ε, πολλούς και διαφορετικούς εταίρους περιγράψαμε την ατζέντα για το 2030 στο κοινό με πολύ απλά λόγια, ότι είναι το σχέδιο για το μέλλον του πλανήτη μας και του κόσμου που κατοικεί σε αυτό. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σχέδιο. Δεν έχουμε έξτρα πλανήτη εφεδρικό, ούτε έχουμε άλλο εφεδρικό πλάνο ή σχέδιο και γι' αυτό είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί πλήρως το σχέδιο αυτό. Από τις έρευνες που έχουμε διεξάγει στην κοινή γνώμη έχουμε δει ότι αυτό το σχέδιο ε, μιλά ξεκάθαρα τη γλώσσα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 25 ετών, διότι αντιλαμβάνονται ότι απευθύνεται στις επόμενες γενιές, τις μελλοντικέ. Είναι ένα σχέδιο το οποίο απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο στους κρατικούς φορείς, αλλά στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, στις επιχειρήσεις, στα πανεπιστήμια, τις ομα... θρησκευτικές ομάδες ή ομάδες πίστης σε οποιονδήποτε έχει όραμα για το μέλλον. Το σχέδιο αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να γίνει στον τομέα της ανάπτυξης ή στον τομέα στον τομέα του περιβάλλοντος. Είναι κάτι που θα εφαρμοστεί και ισχύει για όλους τους τομείς της διακυβέρνησης μιας κοινωνίας. Πώς εξελίσσεται. Έχουμε μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο το έχουν αφομοιώσει τα διάφορα κράτη και είδαμε ότι πάνω από 100 κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να παίρνουν το θέμα πολύ στα σοβαρά. Και μάλιστα ιδιαίτερος ε, σοβαρά παίρνουν το θέμα οι χώρες BRICS πολύ σοβαρά παίρνουν το θέμα πολλές και διαφορετικές χώρες σε διαφορετικές υπήρους. Και ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις το παίρνουν το σχέδιο αυτό στα σοβαρά ε, δείχνει ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος από αυτό που είδαμε με τους στόχους της χιλιετίας. Μάλιστα θα έλεγα ότι μετά από ένα χρόνο η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην αφομοίωση, υιοθέτηση και εφαρμογή αυτού του σχεδίου προσωμιάζει με την πρόοδο των στόχων της χιλιετίας μετά την πάροδο 6 ετών τότε. Σε ένα χρόνο έγιναν γι' αυτό ό,τι δεν είχε γίνει σε έξι χρόνια στο θέμα του στόχων της χιλιετίας και το Σεπτέμβριο αυτής της χρονιάς τελικά εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση. Είδαμε ότι η κοινή γνώμη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το σχέδιο αυτό. Το έχουν μάθει και το έχουν ακούσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι και μέλη των κοινοβουλίων παντού σε όλες τις χώρες το παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Στις συζητήσεις που έχουμε με τη Διακοινοβουλευτική Ένωση αυτό που ακούμε είναι ότι τα μέλη των κοινοβουλίων ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτό το θέμα παρά για οποιοδήποτε άλλο θέμα της ε, ανάπτυξης διεθνώς. Αυτή τη χρονιά προέκυψαν και κάποιοι κινητήριοι μοχλοί ανάπτυξης που όθησαν αυτό το σχέδιο προς τα εμπρός ακόμα περισσότερο. Πρώτον, είχαμε την 21η διάσκεψη των μερών και το αποτέλεσμα αυτής άρχισε να ισχύει πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Είδαμε ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν εκπεφρασμένη βούληση η αφήγηση για το κλίμα και η αφήγηση για την ανάπτυξη να συνδεθούν έτσι ώστε όλες οι δραστηριότητες να έχουν χαμηλό ενεργειακό ενεργειακό αποτύπωμα, να έχουν χαμηλή κατανάλωση άνθρακα και να μπορέσουν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πριν από κάποιες εβδομάδες, δύο μάλλον, στην 22η διάσκεψη των μερών στο Μαρακές, μίλησα με εκπροσώπους κυβερνήσεων και διαπίστωσα ότι για όλους ε, η ανάπτυξη στο μέλλον πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με το κλίμα. Οι κυβερνήσεις παντού στον κόσμο ε, σπρώχουν και ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση για ισότητα στις ευκαιρίες, ε, για αυξημένη πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης και για ε, μείωση των ανισοτήτων, ειδικά των ανισοτήτων που οφείλονται στο φύλλο, κάτι το οποίο ταιριάζει εξαιρετικά με την ατζέντα για το 2030. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η σχέση ε, μεταξύ της ατζέντα αυτής και της μαζικής μετανάστευσης. Στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Υόρκη στις 19 Σεπτεμβρίου είχαμε σύνοδο για τη μετανάστευση και υπήρξαν συμφωνίες για την προσέγγιση του θέματος αυτού με ενδιαφέρον συνολικό γιατί οι προκλήσεις που υψώνονται είναι πολύ μεγάλες στην Ασία, στην Αφρική αλλά και στην Ευρώπη. Επομένως είναι σαφής ο δεσμός μεταξύ των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης και της ανάγκης εφαρμογής της ατζέντα για το 2030. Επειδή η συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα έχει πολύ μεγάλο νόημα για πάρα πολλούς ανθρώπους, θεωρούμε ότι ο καθένας οπουδήποτε θα πρέπει να έχει ρόλο, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και την ιδιότητα και να παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής αλλά και να αποδίδει λογαριασμό αναλόγως για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το σχέδιο αυτό. Είναι εξαιρετικά σημαντική η ενεργή εμπλοκή και συνεισφορά των επιχειρήσεων. Οι ιδιωτικέ επενδύσεις, η ιδιωτική κεφαλαιοχική δράση είναι αυτή που τελικά θα οδηγήσει στην εφαρμογή του σχεδίου με σωστό τρόπο. Όμως η διαφάνεια απαιτεί έλεγχο των οικονομικών, ε, η διαφάνεια απαιτεί λογοδοσία. Αυτά είναι που θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Άρα σε αυτό το σκέλος έρχεται η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών να συμβάλλει. Να σα πω ότι τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών έχουν δεσμευθεί να στηρίξουν την εφαρμογή της ατζέντα για το έτσι ώστε το 40% των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο να είναι σε θέση να την αποκτήσουν έτσι ώστε τουλάχιστον να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της εφαρμογής της ατζέντα αυτής. Να σας πω ποια είναι τα επόμενα βήματα. Μέσα στο σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτή τη στιγμή γίνονται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές για τον τρόπο, στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, δουλεύουμε, επικοινωνούμε, χρηματοδοτούμε τις δραστηριότητε μα και αποδίδουμε λογαριασμό για τα πεπραγμένα μα, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούμε, να ευθυγραμμιστούμε πλήρως με αυτή την απολύτω επαναστατική ατζέντα για εμά. Απαιτεί η ατζέντα αυτή να σκεφτόμαστε και να δουλεύουμε οριζόντια, να υπάρχει ενεργή ε, συνεισφορά και εμπλεκή των πάντων και μάλιστα να επιδεικνύουν όλοι πνεύμα φιλοδοξία έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν τα επιθυμητά τα επιθυμητά αποτελέσματα. Διασφαλίζουμε λοιπόν την με, ε, ομαλή μετάβαση της πολιτικής ηγεσία του, του ΟΗΕ από τον κύριο Μπαν Κιμούν στον κύριο Αντώνιο Γκουτιέρες έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόσκομα ε, ως προς την πορεία του σχεδίου αυτού, της ατζέντα αυτής. Θα είναι οι προκλήσεις πολύ σημαντικές, ειδικά σε ό,τι αφορά το Go14, τη δουλειά για τους ε, ωκεανούς, τη δουλειά για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, αφού χωρίς ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει και ανάπτυξη. Τέλος, ε, παρατηρούμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει αυτές τις ανακοινώσεις και αυτό δείχνει ότι η Ευρώπη και ως κοινωνίες και ως θεσμικά όργανα και ως κρατημέλη και ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, έχει ενεργό ρόλο έτσι ώστε η δουλειά αυτή να χαρακτηρίσει εσύ θέμελα την ίδια την Ευρώπη στη μελλοντική της πορεία. Κάτι το οποίο θα έχει θετικό αντίκτυπο και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Στρέφουμε τώρα προς τους συναδέλφους που θα ήθελα να θέσουν ερωτήσεις. Νέρς πρώτο Πρώτος ομιλητής, παρακαλώ. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ, κύριε Νεμπάρο. Γνωριζόμαστε ήδη. Ήθελα να εστιαστώ στη χρηματοδότηση. Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για το 2030. Τα πρώτα 15 χρόνια των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης έχουμε επιτύχει, και αυτό κάνει έκπληξη, πολλούς από τους στόχους, ε, ειδικότερα ε, υπό τον Κοφιανάν και την αρίστη διαχείρισή του. Ε, και αναρωτιόμουν όσον αφορά τη χρηματοδότηση που θα απαιτηθεί για την επίτευξη των ε, στόχων της ατζέντα του 2030. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας ότι απαιτούνται τεράστια χρηματικά ποσά για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων. Μιλάμε για 3 εκατομμύριο δολάρια. Αναζήτησε λοιπόν νέους τρόπους χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Πρώτα απ' όλα με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και δεύτερον ε, ε, προσαρμόζοντας ε, τα οικονομικά ώστε τα κονδύλια να, να μόχλευση των κονδυλίων και στο πλαίσιο συνεργασιών ε, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και ήθελα να μου πείτε κύριε Ναβαρό πώς προβλέπετε τις απαιτήσει χρηματοδότησης, πώς θα γίνει η χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζητάμε από τους φορολογουμένους να χρηματοδοτούν, θα βρούμε νέου τρόπου χρηματοδότησης, ειδικότερα με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα που έχει πολλά χρήματα. Είναι και κομμάτι της πράσινης οικονομίας. Δεν είναι. Είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι κερδίζουν. Ε, και αν η πράσινη οικονομία ε, αποτελεί κομμάτι μιας ε, πιο οικουμενικής οικονομίας, τότε όλοι κερδίζουν, γιατί με τις νέες τεχνολογίες τεράστιες είναι οι ευκαιρίες που, θα, που υπάρχουν για δημιουργία νέων τεχνολογιών, νέων τρόπων προστασίας του περιβάλλοντος, Δημιουργώντα ταυτόχρονα θέσει εργασία και ανάπτυξη. Τι, έχετε, τι θέση έχετε γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Ε, κύριε Σνόιζερ. Σας ευχαριστώ. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος ε, Τιμάρμανς, μετά από την υιοθέτηση των SDGs ε, το Σεπτέμβριο του 2015 δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι απλά σε, μέσα σε θύλακες περιορισμένα. Θα πρέπει δηλαδή η υιοθέτηση αυτή των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελέσουν μία ευκαιρία προκειμένου να αλλάξουμε όλοι μαζί από κοινού. Και ιδιαίτερα από την οπτική γωνία τη δική μας της Επιτροπής δηλαδή Ανάπτυξης προσπαθούμε να υιοθετήσουμε αυτήν την ε, κατάργηση της διάκρισης ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ανεπτυγμένες χώρες. Όλες είμαστε χώρες οι οποίες αναπτυσσόμαστε και προσπαθούμε να κατευθυνθούμε προς την επίτευξη του στόχους, ε, των στόχων που θέσαμε από καινού έως το 2030. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στα προβλήματα τα οποία καλούμαστε ακόμα να ε, επιλύσουμε και θα έπρεπε να είχαμε επιλύσει έως το 2015, αναφέρομαι δηλαδή στους ε, στόχους της χιλιετίας. Ε, πολλούς από αυτούς τους στόχους τους επιτύχαμε, αλλά κάποιους ε, από αυτούς όχι, οπότε θα πρέπει να συμπεριλάβουμε αυτούς τους στόχους που δεν επιτύχαμε ακόμα στους νέους στόχους έως το 2030. Αυτή λοιπόν η αλλαγή στη σκέψη μας, στην προσέγγιση μας που ανέφερα, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Αλλά εάν προσπαθήσουμε πραγματικά να έχουμε αυτή τη συνέχεια μεταξύ των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας με τους ε, νέους βιώσιμους στόχους σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την αντιμετώπιση της οικονομικής ε, κρίσης θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και από τη μία πλευρά να ασχολούμαστε με επίκαιρα ζητήματα και από την άλλη πλευρά να διατηρήσουμε το όραμα και τους στόχους που σε μακροπρόθεσμο επίπεδο στο 2030. Νομίζω και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της κοινωνικής ε, ένδυας και ε, την προστασία των πόρων από κατασπατάληση ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει ανάπτυξη. Ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι ο Κάλφ Φάλκεμπερκ διορίστηκε ως ειδικό σύμβουλος του Προέδρου της Επιτροπής για αυτό το ζήτημα. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό συνεργάζεται μαζί σας με τα Ηνωμένα Έθνη ο κ. Φάλκεμπερκ. Και από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά τις δύο ανακοινώσεις οι οποίες αναφέρθηκαν, νομίζω πως ε, η έκθεση του Κοινοβουλίου θα οριστικοποιηθεί σε λίγο σε ό,τι αφορά το κοινό σύμφωνο και αυτό νομίζω πως ε, θα μας βοηθήσει να χαράξουμε και, τον, την πορεία που θα ακολουθήσουμε για την επίτευξη των ε, στόχων στο 2030. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μασελές, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να αναφερθώ στα, οικονομικά, στα οικολογικά εγκλήματα, στις ε, πράξεις που επιβαρύνουν τα οικοσυστήματα και κάνουν τους ανθρώπους που ζουν στη συγκεκριμένη επικράτεια να κινδυνεύουν. Μιλούμε για οικολογική γενοκτονία. Είναι ένας άλλος ορισμός των οικολογικών ε, αδικημάτων, οικολογικών εγκλημάτων, ε, για τα οποία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό οι πολυεθνικές εταιρείε με τη καλλιέργεια του φινικέλαιου, των ε, αντίστοιχων δέντρων για την παραγωγή του φινικέλαιου, οδηγούν σε πλήρη αποδάσωση και απερίμωση ε, ολόκληρα δάση στην Αμαλεσία, ε, στην Ινδονησία, πάρα πολλά μέρη στον κόσμο, μεταξύ άλλων. Πώς θα προσεγγίσετε αυτό το θέμα μέσα στο πλαίσιο της ατζέντα του 2030. Δεν μπορεί να υπάρξει ε, ανάπτυξη με οικολογικά εγκλήματα τέτοιου βεληνικούς, τα οποία τελικά ε, κάνουν την ασφάλεια των ανθρώπων να κινδυνεύει. Άρα και την ασφάλεια της επικράτειας της εκάστοτε και άρα την ειρήνη στην συγκεκριμένη περιοχή. Πολύ συχνά έχει γίνει λόγος ε, ε, για το ότι ε, θα πρέπει το πέμπτο έγκλημα κατά της ειρήνης να θεωρηθεί το οικολογικό έγκλημα και να συμπεριληφθεί αυτό στη συνθήκη της Ρώμης. Θα ήθελα να υπάρξει τέτοιου είδους διατύπωση, να μιλήσουμε για οικολογικά εγκλήματα και για τις κυρώσεις αυτών. Πώς πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχέδιο και στην ατζέντα για το 2030. Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών μας έχει ξεπεράσει. Έχουμε το Διεθνές Δικαστήριο το, εναντίον της Μονσάντο που ε, συνεδρίασε πριν από ένα μήνα στη Χάγη. Πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα έτσι ώστε οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να μην τελικά ε, καταφέρονται εναντίον του περιβάλλοντος και της ζωής των μελλοντικών γενναιών. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ κάποιε ερωτήσει τόσο για τον κύριο όσο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει στείλει εδώ εκπροσώπου από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο και την ε, Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ. Πολύ σωστά είπατε κύριε Ναβάρο ότι η πρόοδο ε, που έχει σημειωθεί είναι καλύτερη από ό,τι για του στόχου τη χιλιετία. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαδικασία εντό των Ηνωμένων ε, Εθνών ώστε οι κυβερνήσει να παρακολουθούν την εξέλιξη ένα φόρουμ υψηλού επίπεδου συναντήθηκε τον Ιούλιο και πολλές χώρες ε, αναφέρουν εκεί ε, το βαθμό υλοποίηση. Πώ γίνεται αυτό, είναι προαιρετικό, εθελοντικό, κρατά κάποιο κατάλογο των χωρών ε, ε, στα Ηνωμένα Έθνη. Μπορείτε λοιπόν να μας περιγράψετε διαδικαστικά πώς γίνεται ακριβώς ε, ο έλεγχος των κυβερνήσεων ότι ε, τηρούν ε, την πρόοδο. Και μετά για την Επιτροπή είχαμε τις δύο ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα και πρέπει να ομολογήσω βέβαια αυτή για τι εσωτερικέ πολιτικέ, για την αηφόρο ανάπτυξη. Δεν την κοίταξα. Θα μπορούσε όμω η Γενική Διευθύνση Περιβαλλοντό να εξηγήσει αυτά είναι απλά αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση των στόχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει, θα συλλέξει δεδομένα από τα κράτη-μέλη, να δει ποιε χώρε υλοποιούν του στόχου και πώ. Γιατί, για να είμαι ειλικρινή, μιλώντα σε υπουργού από τη χώρα μου, ο μόνο που συζήτησε, που είχε να πει κάτι, ήταν η ο Υπουργό Ανάπτυξη. Όποιο ασχολείται με την, ο περιβάλλον δεν είχε να πει τίποτα. Πολλοί εκπρόσωποι τη κυβέρνηση δεν είχαν να πούν τίποτα. Θα έπρεπε όμω να εμπλέκονται και οι Υπουργοί Μεταφορών, ε, Γεωργία, ε, δεν βλέπω όμω πολλέ τέτοιε συνδείξει στη δική μου χώρα και αναρωτιέμαι, οι συνάδελφοι εδώ ε, ρωτούν τι κυβερνήσει του τι γίνεται με. Ε, ρωτούν αν, ότι, αν υπάρχει πολιτική συνοχή μεταξύ όλων των ε, Υπουργείων. Εδώ έχουμε την Επιτροπή περιβάλλοντο και Υπερβάλλοντο, αλλά θα έπρεπε να έχουμε και συναδέλφου από την ε, Επιτροπή Αλληλεία, Μεταφορών, Πώς ε, θα τα συντονίσει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το τι κάνουν τα επιμέρους κράτη-μέλη. Μπορούμε να αναμένουμε δηλαδή κάποιε εκθέσει προόδου που θα εμφανίζουν συγκεντρωτικά όλε αυτέ τι πληροφορίε. Δεν βλέπω να ζητούν άλλοι συνάδελφοι τον λόγο, οπότε α το ότι αυτό ήταν ο πρώτο γύρο ερωτήσεων. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Ναμπάρο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ξαναβλέπω τον κύριο Τίβερ και ευχαριστώ για τα σχόλια σας όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Η, χρηματο... η διάσκεψη για τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη που έλαβε χώρα στο Ιωχανέσμπουργκ τον Ιούλιο του 2015 συμπέρανε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια συμβάλλει στην ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης. Αλλά δεν είναι αυτή η κύρια οδός μέσω της οποίας ε, θα χρηματοδοτηθεί αυτή, αυτό το εγχείρημα. Ο βασικός τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθούν ε, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ε, είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα επιδιώκουν όλο και περισσότερο τους ε, στόχους βιοσανάπτυξης ως ένα πλαίσιο εντός του οποίου διεξάγουν ε, τις δραστηριότητές τους. Το πόσο όλα αυτά θα γίνουν ε, φυσικά βασίζεται στην προαιρετική συμμετοχή των επιχειρήσεων αλλά παρατηρείται μια μεγάλη αλλαγή νοοτροπίας τον τελευταίο χρόνο τεράστια αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που μας ενημερώνουν στα Ηνωμένα Έθνη ότι είναι έτοιμες να ελεγχθούν στο πλαίσιο του συνόλου των στόχων ε, ε, βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή στους λογαριασμούς τους, δεν υπολογίζουν μόνο τα χρήματα που έχουν δαπανίσει, αλλά και το διοξίδιο του άνθρακα που, έχουν εκλήσει, που ε, που έχουν κλείσει ε, και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και αυτό αφορά όλους τους τομείς, το τομέα των ορυχείων, τις μεταφορές. Έχουμε λίγη δουλειά ακόμη να κάνουμε με τις θαλάσσιες μεταφορές από ότι με τις εναέριες και τις οδικές μεταφορές, όπου σημειώνεται ήδη πρόοδος. Και επίσης ε, κάποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρήση της γης, όπως η γεωργία και η δασοκομεία. Αλλάζοντας λοιπόν τη φύση των δραστηριοτήτων ώστε να υπάρχει κάποια ε, υπευθυνότητα σε σχέση με τους στόχους βιωσιμής ανάπτυξης. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου επιχειρήσει ουσιαστικά είναι ο βασικός κινητήριος ε, μοχλός ε, για την υλοποίηση των SDG και αυτό ισχύει περισσότερο για τους στόχους που αφορούν αστικά θέματα και υποδομές. Η αναπτυξιακή βοήθεια έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στο να παράσχει κάλυψη κινδύνου για τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε δύσκολες περιοχές αλλά και για τη συγχώνευση των χρηματοδοτήσεων ώστε το ιδιωτικό τομέα να μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα που κανονικά δεν θα έπρατε όπως υπηρεσίες για πολύ φτωχούς ανθρώπους. Κύριε Ντίβερ, να σας πω, ε, έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα οικονομικής καινοτομία, ειδικά σχεδιασμένη για να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για τέτοιου είδους ε, ε, συμμετοχή και θα ήθελα να σας καλέσω να συμμετάσχετε και εσείς για να δείτε ακριβώς πώς γίνονται τα πράγματα και ακούσαμε πολλές ερωτήσεις μετά κύριε Νόιζερ, από σας πολλές ερωτήσεις. Θέλω να σας πω ότι η ηγεσία που επέδειξε ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς ήταν πολύ σημαντική και όπως είπατε αυτός αναγνώρισε τις ευκαιρίες που έχουν πιθανώς να προσφέρουν οι SDGs στους τρόπους λειτουργίας των κυβερνήσεων αλλά και στον τρόπο με τον οποίο όλοι σκεφτόμαστε ώστε να βγούμε από την περιορισμένη σκέψη που πολλοί από εμά πιστεύουμε σήμερα ότι τα περασμένα χρόνια λειτουργήσε ω μειονέκτημα. Να πω ότι στο πλαίσιο των SDG η διαφορά των αναπτυσσόμενων και των ανεπτυγμένων χωρών είναι πλέον λιγότερο σαφή. Θέλουμε μάλιστα να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο ανεπτυγμένε χώρε, διότι έτσι όπω το βλέπουμε εμεί, καμία χώρα δεν είναι ανεπτυγμένη. Όλοι εξακολουθούμε να αναπτυσσόμαστε. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί η υλοποίηση των στόχων ε, των αντιξακτικών στόχων της χιλιετίας, ειδικότερα σε δύσκολους τομείς όπως η υγεία και η παιδεία. Συμφωνούμε μαζί σας ότι η αλλαγή από ένα κατακαιρματισμένο τρόπο εργασίας σε έναν πιο οικουμενικό ολοκληρωμένο τρόπο εργασίας χρειάζεται κάποιο χρόνο και ε, δουλεύουμε εντατικά για αυτό το σκοπό στα Ηνωμένα Έθνη και συνδέονται, ξέρετε, πολύ στενά ζητήματα όπως η προσφυγική κρίση ή κάποιες εμπορικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, και η στοχή ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Ουσιαστικά η πλήρης υλοποίηση των SDG μειώνει τον κίνδυνο ε, προσφυγικής χρήσης και μετανάστευσης. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο και περισσότερο Ευρωπαίοι ηγέτε μου λένε ότι είναι δυνατή η εφαρμογή των SDG στι δικέ του χώρε. Και να πω ότι εμεί στα Ηνωμένα Έθνη συνεργαζόμαστε στενά με επιτρόπου και του εκπροσώπου του ώστε να συνεχιστεί μια ισχυρή ε, δέσμευση και ε, την οποία θα εκφράσουμε μέσα από τις ε, ημέρες που θα φερωθούν στην ανάπτυξη. Να πω κύριε Μαζελέζη, ότι σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και οι συνάδελφοί σας ήταν πολύ σαφείς μαζί μας. Υπάρχουν πολλά που απομένουν να γίνουν για να εστιάσουμε όλο και περισσότερη προσοχή στη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όσον αφορά την περιβαλλοντική καταστροφή και ώστε να βρεθεί κάποιο τρόπο να ε, καλούνται πρώτων ευθυνών του σε τέτοιε περιπτώσει. Γι' αυτό το λόγο η ανακοίνωση με τα βήματα για ένα ε, βιώσιμο μέλλον είναι πολύ σημαντικά. Ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη ε, δεν συμβαίνει μόνο στην Ευρώπη. Έχει επιπτώσει και εξωτερικά. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες ε, προαιρετικές ε, όσον αφορά τη χρήση της γης, την πρόσβαση στα ύδατα μέσω ε, της Επιτροπής για τη Διατροφική Ασφάλεια στη Ρώμη. Υπάρχει μια επιτροπή που εξετάζει τα ζητήματα πρόσβασης στη γη και στα ύδατα και οποιαδήποτε παραβίαση μπορεί να απειλήσει την ειρήνη. Και εμείς συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Πρόκειται για έναν τομέα που χρειάζει προσοχής εμείς εντός των Εθνών βασιζόμαστε στα κράτη-μέλη μας ε, για να προχωρήσουν όλα αυτά με την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Και τώρα να ε, στραφώ στη Λίντα Μακαβέν για την ερώτησή της για το κατά πόσο έχουμε ένα μηχανισμό διασφάλισης του ότι οι κυβερνήσεις παρακολουθούν την πρόοδο. Να σε απαντήσω το εξή. Μιλάμε για ένα σύνολο συμφωνιών που δεν είναι νομοθεσία, βασίζονται στη συνένεση η ευθύνη εφαρμογής αναπόκειται πρωταρχικά στις εθνικές κυβερνήσεις από τις οποίες ε, αναμένουμε να παρακολουθούν την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέσω διαδικασιών εντός των χωρών ε, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και άλλων τμήματων της κοινωνίας αλλά εντός των Ηνωμένων Εθνών μέσω του ε, ε, Υψηλού Πολιτικού Φόρουμ και άλλων μηχανισμών σίγουρα θα ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές και θα ε, δημοσιοποιούμε ό,τι παρατηρούμε να γίνεται στις χώρες σε θέματα διαφάνειας και ευθύνης. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στην παρακολούθηση της πρόοδου των στόχων αυτής της ατζέντα. Δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη και το περιβάλλον, αφορά όλους τους τομείς. Εμεί αυτή τη στιγμή έχουμε μια σύνοδο κορυφή στο Ασκαμπάτ ε, για τις βιώσιμε μεταφορές ε, και φυσικά θα έπρεπε να συμμετάξει αυτή η Επιτροπή Μεταφορών. Ο τομέα τη γεωργία, ο τομέα τη Υγεία. Ε, είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο της ανθρωπότητας ολόκληρη. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων λοιπόν και το Συμβούλιο επίση θα έπρεπε να συμμετέχουν. Πρέπει όλοι μας ε, να μεριμνήσουμε ώστε το ζήτημα αυτό να εξετάζεται από ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν ε, ότι θα βοηθήσουν μάλιστα και για αυτό το σκοπό και οι συναδέλφοι από την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν βλέπω ότι ζητούν το λόγο και άλλοι συναδέλφοι. Βλέπω ότι είναι συναδέλφοι από την Επιτροπή Περιβαλλόντος και θέλουν να, ζητήσουν, να κάνουν ερωτήσει. Βλέπω την κυρία Μυρία Μτάλη. Δεν βλέπω το όνομά σας, παρακαλώ. Και η κυρία Σερία Φιρίκ. Κάποιο άλλο συνάδελφο που θα ήθελε να κάνει ερωτήσει. Ωραία, α ακούσουμε αυτούς τους, ε, τα, αυτά τα δύο μέλη και μετά θα ακούσουμε την Κομισιόν. Θα ήθελα να θέσω ε, δύο ερωτήματα και εγώ σε σχέση με προηγούμενα ερωτήματα που τέθηκαν, αλλά και σχέση με μια δήλωση που κάνετε τώρα, γιατί είπατε ότι θα πρέπει ε, και οι κυβερνήσεων και γενικά οι να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Και ένα από τα σημεία κριτική ε, που αναφέρθηκε είναι ότι σε αντίθεση με του ε, στόχου MTG οι SDGs δεν επιτρέπουν να εστιάσουμε τόσο πολύ σε περιφερειακό επίπεδο. Αν συμφωνείτε λοιπόν με αυτή την αξιολόγηση ε, τότε δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι και στο μικρό επίπεδο, δηλαδή σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο είναι σημαντικό να γίνουν προσπάθειες για να ανταποκριθούμε ε, σε αυτούς τους στόχους και κατά συνέπεια ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις εθνικές ιδιαιτερότητες. Με άλλα λόγια, πώς τα Ηνωμένα Έθνη θα διασφαλίσουν ότι θα ληφθεί αυτή η διάσταση υπόψη τους ώστε να, να εφαρμοστούν στην πράξη αυτή οι στόχοι. Μετά, αναφερθήκατε και στην σημασία του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη αυτών των στόχων αλλά κάποια διεθνή μέσα ανέφεραν ότι 2 ε, 3 ε, ε, ευρώ σε επίπεδο δηλαδή κρατικών χρηματοδοτήσεων θα χρειαστούν έως το 2030, δηλαδή γύρω στο 4% του ΑΕΠΑ, των λόγων χώρων. Ε, ταυτόχρονα όμως οι δεσμεύσει από την πλευρά της, ε, των ενισχύσεων της βοήθειας των κρατών είναι της τάξης του 0,7%. Οπότε πώς θα καλύψετε αυτό το έλλειμμα της χρηματοδότησης. Ε, ευχαριστώ κύριε Πεπέ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά γιατί δεν είναι δυστυχώς, δεν έχω διερμηνία από τα Ολλανδικά. Ε, ε, ε συμφωνώ και με τον ε, πρόεδρο τη Επιτροπή δηλαδή, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και να συμφωνήσουμε επί συγκεκριμένων ζητημάτων και με την Επιτροπή Γεωργία. Γιατί μία σειρά από αυτά τα ζητήματα συζητώνται και θα πρέπει να εφαρμοστούν ακριβώ στο γεωργικό τομέα. Έχουμε δηλαδή τον. Ε, ζήτημα που, που έχουν ε, αναφέρει επανειλημμένα οι συνάδελφοι σε ό,τι αφορά την κοινοτομία, το σχέδιο Juncker ε, και από εκεί και μετά θα πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε ή όχι. Να συμφωνήσουμε δηλαδή μεταξύ μας. Είναι ένα σημαντικό αυτό το ζήτημα. Και θα πρέπει να συζητηθεί και μεταξύ μας εδώ, δηλαδή μεταξύ των διαφορετικών επιτροπών. Και βλέπω εδώ και τον κύριο Λαβία Και ε, πραγματικά θα πρέπει να ξεκινήσει ένας ε, διάλογος ε, σε αυτό το επίπεδο, όχι μόνο για τις υπόλοιπε χώρες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να γίνει και μεταξύ των πολιτών, δηλαδή στο επίπεδο της κοινωνία των πολιτών να ξεκινήσει ο διάλογος. Ελπίζω να με καταλάβατε σε αυτά που ανέφερα. Ευχαριστούμε, λέει πρόεδρο. δεν βλέπω κάποιο άλλους συνάδελφου να ζητάει το λόγο, οπότε θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή, γιατί τέθηκαν κάποια ερωτήματα και προ την Επιτροπή και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Νεμπάρα. Κύριε Τιμοβίκη, νομίζω εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο από την Επιτροπή. Α, είστε εκεί, παρακαλώ. Ε, και συστηθείτε αν θέλετε. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλου. Δημοβίλη λέγομαι, ε, εργάζομαι για τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ε, από την Επιτροπή. και ε, εγώ ασχολούμαι ιδιαίτερα με το ζήτημα των στόχων SDG και με τα θέματα που περιέγραψε τόσο λαφρά ο κύριος Ναμπάρο, δηλαδή αυτή την ε, δύσκολη διαδικασία του σχεδιασμού των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Τώρα βέβαια κινούμαστε προς τη φάση της εφαρμογής των λόγων στόχων, οπότε να ευχαριστήσω καταρχήν ε, τον κύριο Ναβάρο για τα ενθαρρυντικά του λόγια σε ό,τι αφορά το λόγο πακέτο και σας ευχαριστώ όλους βέβαια και για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει και για τα ερωτήματα δηλαδή που θέσατε από την πλευρά των Προέδρων, των Επιτροπών και των Μενών. Ε, νομίζω πως ε, δεν μπορούμε τώρα σήμερα να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες ε, αυτού του πακέτου. Θα μας δοθούν διάφορες ευκαιρίες για να το κάνουμε, δηλαδή και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου. Αλλά επιτρέψτε μου να αναφέρω, να θίξω ένα-δυο ζητήματα που τέθηκαν σήμερα και από ε, του συναδέλφου και από τον κύριο Ναμπάρο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν έχει διαθετήσει ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη που αναφερόταν ήδη στην ε, συνθήκη του Άμστερνταμ και γενικότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη ως μέρο δηλαδή των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και από το 2001 έχουμε την ε, στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ από το 2010 έχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη ως ένα μέρος που έχει ενταχθεί σε όλες τις πολιτικές ε, της Ένωσης, όπως για παράδειγμα για την ε, στρατηγική 2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτελέσει κινητήρια δύναμη, αν θέλετε, ε, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του θεματολογίου της ατζέντα του 2030 και επιθυμούμε προφανώς να στεφτεί με επιτυχία τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε δηλαδή να εφαρμοστούν επιτυχώς οι στόχοι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη έχουν γίνει μια σειρά από αλλαγέ στο πακέτο το οποίο θέτησε η Επιτροπή ε, πέρυσι, οπότε δεν θα επισέλθω στα επιμέρου στοιχεία αυτού του πακέτου. Απλώ επιτρέψτε μου να πω ότι ε, αν δούμε αυτό το πακέτο θα διαπιστώσουμε ότι με βάση την παράδοση που έχουμε στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης ως Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούμε από ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας αν θέλετε ήδη έχει κατοχυρωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα ε, διαπιστώνουμε σε αυτό το πακέτο ότι θα πρέπει να ε, δώσουμε ακόμα περισσότερη έμφαση, να υποστηρίξουμε αυτές τις πολιτικές κατά το σχεδιασμό των ε, περαιτέρω σχεδίων των περαιτέρω πολιτικών. Η απάντηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το πώς ανταποκρίνεται, αν θέλετε, ε, στην επίτευξη αυτού του θεματολογίου του 2030 και αυτό το λέω για όσους δεν έχει διαβάσει τη σχετική ανακοίνωση ε, έχει δύο κύριους άξονες από τη μία πλευρά έχουμε ε, την ευθυγράμμιση με τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την άλλη πλευρά έχουμε την ευθυγράμμιση των πολιτικών μας και την εφαρμογή αυτών των πολιτικών στις διάφορες θεματικές τομεακές ε, πολιτικές ακριβώς προκειμένου να προσανατολίζονται στους στόχους ε, SDGs. Ε, σε ό,τι αφορά την συνεκτικότητα των σχετικών πολιτικών, το ζήτημα που αναφέρθηκε, προφανώ το αναγνωρίζουμε ότι είναι ανάγκη να υπάρχει συνοχή των σχετικών πολιτικών και χρειάζεται κατάλληλη πληροφόρηση και εδώ στο Κοινοβούλιο και χρειάζεται και συνεργασία μεταξύ όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών της ε, Επιτροπής, ε, τόσο στο επίπεδο της ε, εφαρμογής και σε ό,τι αφορά ειδικότερα την σχεδίαση των εφαρμοστικών μέτρων αυτών των στόχων σε επίπεδο της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο τώρα της διακυβέρνησης, σε επίπεδο Επιτροπής, θα ευθυγραμμίσουμε, θα εντάξουμε δηλαδή τις πολιτικές, στις πολιτικές και στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτούς τους στόχους ως βασική αρχή και συγκεκριμένα ε, με τους εξής τρόπους. Θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα ε, εργαλεία νομοθεσίας, νόμο παραγωγής, ούτως ώστε να εντάσσονται σε αυτές τις πολιτικές συνέσεις. Όχι. Επίσης θα λαμβάνουμε υπόψη μας τις τρεις διαστάσεις, δηλαδή την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική, με ισορροπημένο τρόπο και από εκεί και μετά σε επίπεδο δομής ο Πρόεδρος μαζί με τους ε, επιτρόπους και το σχετική το σχετικό συμβούλιο ε, των επιτρόπων που έχει σχηματιστεί αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο ε, για την εργασία σε αυτό το ε, τομέα και προκειμένου ακριβώς να υπερκεράσουμε αυτή την κατακαιρματισμένη προσέγγιση σε επίπεδο πολιτικών που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα. Ο αντιπρόεδρος Τίμερμαν θα παίξει έναν συντονιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του συνόλου τη Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, την πρόοδο εφαρμογή των στόχων τη Ατζέντα 2030. τέθηκε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά το monitoring, την παρακολούθηση δηλαδή του της εφαρμογής, της προόδου της εφαρμογής των στόχων. Επιτρέψτε να πω ότι όταν η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της, το σκεπτικό της ήταν ότι οι SDGs αποτελούν μια ατζέντα συνεργασίας, ε, δηλαδή ε, και οι κυβερνήσεις ε, και όλοι οι δημόσιοι αλλά και μη κυβερνητικοί φορείς θα συμμετάσχουν εδώ και η παρακολούθηση της εφαρμογής λοιπόν θα λάβει χώρα από κοινού, από όλου αυτού του ε, φορέ. Ε, η ανακοίνωση αποτελεί ένα πλαίσιο εφαρμογή, ακριβώ δίνει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή ε, στα κράτη-μέλη και ένα, μια σειρά από τα οποία ακριβώ αποτελούν τροχοπέδι για την βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο κρατών μελών. Και τα ίδια κράτη-μέλη βρίσκονται ακριβώ αυτή την περίοδο στη φάση σχεδιασμού των δικών του συνέδρων σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη. Όπω είδαμε και στο περσινό φόρουμ ε, υψηλού επίπεδου σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, είδαμε ότι πολλά κράτη-μέλη πράγματι είχαν ανακοινώσει την προετοιμασία των δικών του ε, σχεδίων. Είναι σημαντικό οι ε, εν λόγω δράσει να ξεκινήσουν εγκαίρω και αποτελεσματικά, ούτω ώστε να επιτύχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Πώ θα διασφαλίσουμε τώρα την εφαρμογή. Ένα γενικό πλαίσιο αναφέρεται ήδη στο πακέτο των ανακοινώσεων και αποτελεί προτεραιότητα του να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πρόοδο και με συστηματικό και διαφανή τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ε, συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα παίξει κεντρικό ρόλο προκειμένου να ε, μεγιστοποιηθεί η ε, εφαρμογή των στόχων και προκειμένου να υπάρχει βέβαια και ανάληψη των ευθυνών απέναντι στους πολίτες και προκειμένου κανείς να μην έχει καθυστερήσεις. Ε, και τα κράτη-μέλη ερωτήθηκαν, ε, ζητήθηκε από αυτά ε, πέρυσι από τον Έθνη να δημιουργήσουν μηχανισμούς για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση προόδου και η Επιτροπή θα αναλάβει ακριβώς αυτή την παρακολούθηση στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Στην σχετική ανακοίνωση, η οποία αναφέρθηκε, δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με τις ανακοινώσεις, σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση συγκεκριμένων δεκτών. Ε, θα υπάρξει ένα πλαίσιο δικτών παρακολούθηση ε, αξιολόγηση επιδόσεων, ε, στην οποία θα συμμετέχουν όλε οι σχετικέ αρμόδιε αρχέ τη Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή επίση θα αναλάβει την υποβολή εκθέσεων σε ό,τι αφορά την πρόοδο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο ε, φόρουμ υψηλού επίπεδου ε, σε παγκόσμιο λοιπόν επίπεδο, πράγμα το οποίο νομίζω πω ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κύριο Ναπάνο. Ε, αλλά όπως σας είπα θα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε πιο εντελώς αυτά τα ζητήματα ε, ε, και με τα μέλη του Κοινοβουλίου σε άλλα φορά, αλλά ενδεχομένω να δώσουμε το λόγο και στον συνάδελφο από την ΔΕΦΚΟ για να σχολιάσει εκείνος ο Σένα Ναμπάρο θα πρέπει να αποχωρήσει νομίζω ε, στις 4, οπότε καλύτερα να ακούσουμε τον κύριο Λίβερ, μετά τον κύριο Ναμπάρο και μετά τον εκπρόσωπο της ΔΕΦΚΟ. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός στη Νέα Υόρκη για τις διεθνείς συνεργασίες για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Θα ρωτήσω τους συντονιστές μου εδώ Μήπως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι αντίστοιχο ή εν πάση μια διάσκεψη, ένα συνέδριο και στρέφομαι και στους συναδέλφους από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητώντας τη βοήθειά τους. Μπορούμε να έχουμε μια παγκόσμια διάσκεψη για το πώς θα εμπλακεί ο ιδιωτικός τομέας στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Μιλούμε για ένα τρεις δολάρια χρηματοδότηση και αυτό δεν είναι αμεληταίο. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη μόχλευση των κονδυλίων. Αυτό έχει υπάρξει πλέον στην νομοθεσία και μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία στο ιστορικό υπόβαθρο. Ο κύριος Ναβάρο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι αμέσως στην ερώτηση της κυρίας Τάλη για να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χρηματοδοτηθεί αυτό το εγχείρημα είναι η επένδυση όλων των δυνατών κονδυλίων. Είτε προέρχονται από κυβερνήσεις, είτε προέρχονται από τις επιχειρήσεις. Κάθε είδους επένδυση πρέπει να συνάδει με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και έτσι θα οικοδομήσουμε ένα μέλλον προς όφελος των λαών. Εάν το κάνουμε αυτό με κρατικά χρήματα μόνο δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Και χαίρομαι γιατί μπορώ να ε, δώσω συνέχεια, όπως είπε και ο κύριος Ντίβα, να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια της συζήτησης και θα μεταφέρω αυτό το μήνυμα αύριο όταν επιστρέψω στη Νέα Υόρκη. Ε, κυρία Ντάλη, αναφερθήκατε και σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπατε ότι α, όλα αυτά πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη το συγκείμενο κάθε φορά, το πλαίσιο κάθε φορά. Και συμφωνώ απολύτως. Η εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο είναι μια εφαρμογή που δεν θα δουλέψει ακολουθώντας μόνο ε, το παγκόσμιο ε, σετ οδηγιών. Ε, πρέπει να εμπλακούν οι τοπικές αρχές και θέλουμε τελικά όλα αυτά να φτάσουν σε τοπικό επίπεδο, να συνεργαστούμε με τους Δήμους, με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση για να λειτουργήσει αυτό το εγχείρημα. Στη κυρία Περέκ, βλέπω ότι υπάρχει Ολλανδική καμπίνα και εσείς δεν μιλήσατε Ολλανδικά. Ε, σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας. Εγώ θα ήθελα όλο το Κοινοβούλιο να εμπλακεί στην παρακολούθηση. Μία Πανκοινοβουλευτική Επιτροπή, η Επιτροπή που εστιάζεται στην ατζέντα για την βιώσιμη ή αηφόρο ανάπτυξη και εξετάζει όλους τους τομείς αυτής. Ε, τώρα μόνο μέρος του Κοινοβουλίου έχει εμπλακεί. Θα μου άρεσε αυτή η συνολική προσέγγιση. Ειδικότερα όταν προσφέρουμε στην ιδιωτική χρηματοδότηση για να πετύχουμε αποτελέσματα. Αλλά συμφωνώ πολύ τους μαζί σας, ο γεωργικός τομέας πρέπει να ε, συμμετάσχει ενεργά. Σας ευχαριστώ και σας αποχαιρετώ αν με απελευθερώνετε. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Πράγματι μπορούμε να απελευθερώσουμε τον κύριο Ναβάρο. Καλή σας επιστροφή και καλό ταξίδι. Θα ακούσουμε όμως και την άποψη της Γενικής Διεύθυνσης Επιτροπής. Εσάς σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Δίνω το λόγο στην ε, Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με λένε Παύλος Γουρό και εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να αναφέρω δύο στοιχεία. Μετά τα σχόλιά σας, κύριε Μακεβάν, για, για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώς το λέτε, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παραμβαίνω. Αύριο ο Επίτροπος Μίμητσα έρχεται εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας εξηγήσει. Και η κυρία Μογκερίνη είχε έρθει τις προάλλες και μίλησε σχετικά. Θέλω όμως εγώ να σχολιάσω αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Η συζήτηση έρχεται σε μια πολύ κατάλληλη χρονική συγκαιρία. Σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων η πρωτοβουλία έτυχε ευρεία στήριξη και αυτό δείχνει ότι τα κράτη-μέλη την εστερνίζονται απολύτω. Ένα από τα θετικά στοιχεία, τα ατού τη συνένεση είναι το γεγονός ότι έχουμε κοινή δήλωση ε, στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη-μέλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στα ε, κράτη και ατομικά αλλά και συλλογικά να προσχωρήσουν σε αυτό το εγχείρημα και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Αυτά λοιπόν από πλευράς ανάπτυξης και εξωτερικού σκέλους της εξωτερικής πολιτικής. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα εμπνεύσουν για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε σε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Να πω δύο λόγια για τη συνένεση για όσους απουσιάζουν αύριο και δεν θα ακούσουν τον Επίτροπο. Βασικός στόχος είναι να έχουμε ένα νέο όραμα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει η συνένεση και αυτό το όρομα να το προσαρμόσουμε στην πολιτική μας, στη νέα ατζέντα, στις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της ευρύτερης, ε, της ευρύτερης παγκόσμιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο προήμιο της ατζέντα μιλούμε ε, για το λαό, το πλανήτη, την ευμερία, την ειρήνη, την εταιρική σχέση. Όλ, αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά. Πίεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά, για να υπάρχουν συνδέσεις για τις τρεις διαστάσεις, για το δεσμό μεταξύ της ανάπτυξης και άλλων πολιτικών ε, που ενισχύουν τη συνοχή. Ένα από τα βασικά μηνύματα της συνένεσης είναι ακριβώς αυτό, ότι θα συνεργαστούμε πιο στενά με τα κρατημέλη στο εκάστοτε αρχηγείο, στην έδρα, επιτόπου για οργάνωση κοινών δράσεων και για συνολική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται αυτό το εγχείρημα για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για την αναπτυξιακή βοήθεια και για να υπάρχει συνολική προσέγγιση κινητοποίησης ιδιωτικών εγχώριων πόρων την ε, βοήθεια θα την επικεντρώσουμε στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες βέβαια θα πρέπει όμως να συνεργαστούμε με τις πιο προηγμένες χώρες για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Αυτά εν συντομία και συνοπτικά για να πω ότι με πολύ μεγάλη χαρά θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ώψη συμφωνίας ή δυνατόν την επόμενη χρονιά και θα έχουμε σημαντικές ευκαιρίες για να τα οριστικοποιήσουμε όλα αυτά. Τις ε, Ευρωπαϊκές ημέρες για την ανάπτυξη πριν, το σχετικό πολιτικό φόρουμ. Νομίζω ότι ο κύριος ε, Ναβάρο ε, επίσης πέτυχε ένα πολύ σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ της συμπληρωματικότητας και του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά για το πώς δουλεύουμε μεταξύ μας οι δύο επιτροπές, αλλά και με τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε, όταν ακούω λόγια τύπου όλοι έχουν ευθύνη, ανησυχώ γιατί τελικά κανείς δεν θα την έχει. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δικές μας κυβερνήσεις είναι υπεύθυνε. Ίσως οι δικοί σας υπουργοί αναλαμβάνουν αυτές τις ευθύνε, αλλά όχι στη δική μου χώρα. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να μην είναι ε, όλα αυτά μόνο όμορφα λόγια διατυπωμένα επί χάρτου στην εκάστοτε σύνοδο του ΟΗΕ. Για να έχει μέλλον ο πλανήτη μας πρέπει όλα αυτά να τα καταφέρουμε. Κύριε Ραβιέρ, έχετε τελικά σχόλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΔΕΒΕ που οργάνωσε αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και για τη φιλοξενία σας. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και οι συναδελφοί μου θα πρέπει να αναχωρήσουμε διότι έχουμε μία συνάντηση σε λίγα λεπτά. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ώστε να αναχωρήσουν οι συναδέλφοι της Επιτροπής Περιβάλλοντος και θα συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ευχαριστώ.